We start voting. Αρχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Audi, the floor is yours. Κύριε Οντή, έχετε το λόγο. Διαδικαστικό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρέμβω με βάση το άρθρο 40, 146 και 148 του εσωτερικού μας κανονισμού. Ε, τη, μιλάμε για, τον, για την πολυγλωσία και την κατάπτωση της ε, πολυγλωσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τροπολογίες 19 έως 28 στις 12 και 40 δεν είχαμε μεταφραστεί στα γαλλικά. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση τη πολυγλωσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό παίρνω το λόγο, για να σε πιστήσω την προσοχή σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, θα το λάβουμε υπόψη μα αυτό στο μέλλον και θα προσπαθήσουμε να επαγρυπνούμε, ούτω ώστε να έχετε εγκαίρω τι μεταφράσει. Τώρα, θα ψηφίσουμε με την απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Μπέγκε για το εργαλείο ευελιξίας. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε με ειδική πλειοψηφία. Τα τρία πέμπτα. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Συγχαίρω τον κύριο Μπέγκε, τον εισηγητή μας. Και τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειές σας κατά την προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Τώρα θα ψηφίσουμε το Γενικό Προϋπολογισμό του 2011. Πρώτη τροπολογία. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Έναρξη. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 21. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ο κύριος Σούλτς θα ήθελε να μιλήσει. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω την εξή εξήγηση για την αιτιολογική η τροπολογία 13. Ο συνάδελφος ε, Γιώργο Φέρμ ε, έθεσε την ε, τροπολογία αυτή στην Επιτροπή. Ε, δεν την ξαναυποβάλαμε, αλλά οι πράσινοι με 40 υπογραφές ε, την ε, επανυπέβαλαν. Θα θέλαμε να απόσχουμε από την τροπολογία αυτή. Έχουμε συμφωνήσει με τους πράσινους στο θέμα αυτό. Ως προς ε, το θέμα συμφωνούμε απόλυτα. Απλά συμφωνήσαμε ότι ως ε, ομάδα δεν θα επανυποβάλουμε τροπολογία, αλλά θα ήθελα να πω ότι ε, στηρίζουμε την φορολογία των οικονομικών συναλλαγών και ελπίζουμε οι συνάδελφοι και από την άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου να μας υποστηρίξουν τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 13. Με ονομαστική ψηφοφορία, εξ ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε όλες τις τροπολογίες ε, στη θέση του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Στην παράγραφο 2 του ψηφίσματος, στην οποία θα ψηφίσουμε πάρα αυτά, θα διαγράψουμε τη φράση υπό την τροποποιημένη της εκδοχή όταν ψηφίσουμε τον προπολογισμό του 2011. Γιατί δεν άλλαξε τίποτα, μια και απορρίψαμε όλες τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Τώρα, θέτω σε ψήφιση το ψήφισμα, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί αν το επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Διαδικαστικό. Η κυρία Ιντζογεύσκα για διαδικαστικό θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να δώσω μια εξήγηση στους συναδέλφους μου. Ψηφίζουμε χωρίς αλλαγές ε, στο σχέδιο που μας παρουσίασε το Συμβούλιο, γιατί είναι επανομοιότυπο με την γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά από εννέα μήνες διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όλους τους εισηγητές. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου και πιστεύω ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε τον προϋπολογισμό του 2011 για να εφαρμοστεί από Πρώτου 2011. Πολύ ωραία, κυρίε και κύριοι. Υιοθετήσαμε τον προπολογισμό χωρί ε, τροπολογίες Όλε οι τροπολογίε απορρίφθηκαν. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα την έκθεση της κυρίας Γεντζογεύσκα. για τον Γενικό Προπολογισμό του 2011. Όλα τα τμήματα του προπολογισμού. Τροπολογίες 2 και 4. Με ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να το τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει πάλι να το τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι πρέπει να το τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα το συνολικό κείμενο. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε το ψήφισμα. Έναρξη της ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε το κείμενο. Συγχαίρω και την κυρία Γεντζογεύσκα και την κυρία Τρούπελ και τις δύο εισηγήτριες. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το Κοινοβούλιο μόλι ανέκρινε τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2011 χωρί τροπολογίε. Φυσικά, εν ονόματι του Συμβουλίου μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την κοινή μα συμφωνία για το προπολογισμό του 2011. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. E, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ακούσετε μια δήλωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε τη διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πέρυσι χρησιμοποίησαμε την απλουστευμένη διαδικασία. Τώρα εφαρμόσαμε τη διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να κάνω την, Ευρωπαϊ... την εξή δήλωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την ε, θέση του Συμβουλίου από τις 10 Δεκεμβρίου του 2010 ε, για το πρόγραμμα προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο. Η δημοσιονομική διαδικασία ολοκληρώθηκε λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης.